certains d'entre vous qui ont envie de prendre la parole pour dire j'ai quelque chose à dire maintenant. Oui. I think another point that came from our group is the linking between generations and that we have an opportunity here to make full use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 auditing every year to share their views on how they treat youth unemployment in a in a sustainable way, not just sustainability when it comes to the environment, but also social sustainability and how they work on youth unemployment. Alors, maintenant, vous avez tous ces deux documents. Je vais vous expliquer comment on va essayer de fonctionner. Donc, vous avez d'un côté un document qui commence par Entering the Labour Market. Celui-là,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

on tienne compte du handicap, on tienne compte de différentes choses et on tienne compte de l'emploi des jeunes. C'est ça votre idée Is it your idea Am I correct Indeed, I want youth employment added to corporate social responsibility, but in the current declaration, I don't see anywhere else where to put it, except under entrepreneurship. Okay. Um,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 companies to provide training and to be recognised for the fact that they are doing that for young people. I don't think it is imposing regulations, it's actually providing them with an opportunity to market themselves even better. Ok, on va arrêter là. Je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour que vous puissiez voter. Donc, dès lors qu'il ne s'agit pas de quotas, etc., mais sur l'idée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 Oui, monsieur. Καλημέρα. Καλημέρα. Ε, σε συνέχεια τον, ε, στο σχόλιο ε, για το συγκεκριμένο θέμα της... Ε, is there a Greek translation? Good. Ε, σε συνέχεια της, ε, της, του σχολείου της Γερμανίδας συναδέλφου για το, για το ε, τρίτο θέμα το οποίο ε, για το οποίο μιλούμε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να προσθέσω ε, κάποια σημεία τα οποία ε, ήρθαν στην εντύπωσή μου μέσω της, της, σελίδας, της επίσημης σελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Facebook, την οποία έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή και κάποια σχόλια τα οποία έχουν γραφτεί εκεί και θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικά και πρέπει να, να υποθούν για την απόψη των νέων οι οποίοι είναι εκεί έξω αυτή τη στιγμή και όντως έχουν μπροστά τους αυτές τις δυσκολίες ε, ε, ένα από αυτά τα σχόλια ε, αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή. τα πιο σημαντικά, εντάξει κάποια ήταν αρκετά έντονα σχόλια, θα τα δείτε και μόνοι σας, αλλά τα πιο σημαντικά έλεγαν για να σταματήσουν τα μέτρα λιτότητα ή τουλάχιστον να συζητήσουμε για τα μέτρα λιτότητα τα οποία υπάρχουν σε αρκετέ χώρε, ε, ειδικά τη Μεσογείου. Ε, Επίση, να σταματήσει η άσκοπη χρήση τη διαδικτυακή προώθηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ε, αυτό δεν δουλεύει πλέον και ε, να, να, να επανεξεταστεί ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αρκετά σχόλια έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σπαταλά ε, πολύ περισσότερα ε, χρήματα από αυτά που χρειάζεται να, να σπαταλήσει. Ε, επίσης, μεγαλύτερος έλεγχος των συνόρων ε, για καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, έτσι ώστε να αποφύγουμε την cheap labor, I don't know that in Greek, το οποίο μεταφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παίρνει ίσως τις δουλειές των νέων ε, και συγκεκριμένα το σχόλιο αυτό ε, που ήθελα να κάνω είναι ε, να σταματήσει η συνεχής αύξηση της, της ηλικίας αφιπηρέτησης. Δηλαδή χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι η ηλικία αφιπηρέτησης ανεβαίνει έτσι ώστε οι νέοι δεν έχουν όσες ευκαιρίες θα μπορούσαν να έχουν στην εργασία αφού οι ήδη υπάρχοντες στην εργασία μένουν για περισσότερα χρόνια.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 À 28, bien sûr. Peut-être à 29, même 30. Ok. Bitte Sie wollen etwas sagen. Thank you. On the very same point, we need, of course, and I very much agree with my French colleague, we need to agree 0.2, 0.5% of what, you know